το λόγο. Thank you, President, and good morning, everyone. Ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Ζητώ συγγνώμη, ξέρω ότι ήταν δύσκολη απόφαση, αλλά ήθελα να πω σήμερα ότι η απόφαση για καθυστέρηση της ψηφοφορίας για τη δικιά μας τουλάχιστον αντιπροσωπεία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή πώς το εκλαμβάνουν οι πολίτες της Ευρώπης. Η ανησυχία μας είναι μεγάλη για αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να το πω και να το τονίσω αυτό. Επίσης... Θα σας δώσω το λόγο μετά τις ανακοινώσεις. Μικρόφωνο παρακαλώ. I have another και έχω και κάτι άλλο για την τροπολογία 27 και η σειρά με την οποία είναι στην ημερήσια διάταξη, γιατί δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες. Θα έπρεπε να την εξετάσουμε συνολικά και το άλλο τμήμα πρέπει να καταπέσει. Συμφωνώ ότι είναι διαδικαστικό, αλλά υπήρξε μεγάλη στήριξη στην τροπολογία 27 και ζητώ από τον Πρόεδρο να το ξανασκεφτεί αυτό το θέμα στο μέλλον. Ακούστε με δύο λεπτά, ακούστε τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου και μετά θα μας πείτε αυτό που θέλετε. Κάποιοι επικεφαλής ομάδων, αρχηγοί ομάδων που εκπροσωπούν την πλειοψηφία στην διάσκεψη των Πρόεδρων ενημέρωσαν τον Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι επιθυμούν να αναβληθεί η ψήφιση της έκθεσης του κ. Λάγκε για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την διατλαντική εταιρική σχέση για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο βάσει πρόταση του Προέδρου, προκειμένου να τροποποιηθεί η μερίσια διάταξη βάση του άρθρου 152. Για να επιτρέψουμε στο Κοινοβούλιο να ψηφίσει αυτή την πρόταση αλλαγή, ο πρόεδρο την αποδέχτηκε. Την υποβάλλει. Έτσι λοιπόν θα ψήφιση την πρόταση αναβολής της έκθεσης Λάγκε για ονομαστική ψηφοφορία. Εάν θέλει κάποιο να μιλήσει υπέρ τη αναβολής και κάποιος δύο λεπτά ένας υπέρ τη αναβολής και ένας κατά. Ποιο θέλει το λόγο υπέρ τη αναβολής εφόσον η πρόταση έχει υποβληθεί επισήμως. Νομίζω πρέπει να σεβαστούμε την βούληση του Κοινοβουλίου. Εφόσον το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει, η αίθουσα μόνο, η Ολομέλεια μόνο έχει την ε, εξουσιοδότηση να αποφασίσει. Η Ολομέλεια αποφασίζει. Παρακαλώ. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, εμείς εδώ και πολλές εβδομάδες προετοιμαστήκαμε για τη σημερινή συζήτηση και τη ψηφοφορία και μάθαμε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί σήμερα η ψηφοφορία. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλέ φήμε. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η δική μα πολιτική ομάδα θα ήταν διατεθειμένη να ψηφίσει σήμερα, αλλά μια και δεν θα διεξαχθεί σήμερα η ψηφοφορία και η Επιτροπή θα πρέπει ωστόσο να ψηφίσει τι τροπολογίε, θεωρούμε ότι έχει νόημα η ψηφοφορία και η συζήτηση να διεξαχθούν από κοινού και στη συνέχεια να ε, συζητήσουμε όταν ξέρουμε τι ακριβώς θα τεθεί στην ε, ψηφοφορία. Άρα λοιπόν διεξαχθεί η ψηφοφορία εφόσον έχουν συνεδριάσει οι, επιτροπές. Παρακαλούμε λοιπόν να αναβληθεί η ψηφοφορία και η συζήτηση. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί κατά της να Αξιότιμοι συνάδελφοι, προηγουμένω στην αιτιολόγηση ελέγχθη ότι η πλειονότητα ή η επικεφαλής των πολιτικών ομάδων έχουν, ε, ε, απευθύνθηκαν προς τον Πρόεδρο ούτως ώστε να μην γίνει σήμερα συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά προβληματική γιατί με τον τρόπο αυτό τελικά θέτουν ένα αμφιβόλο και ακυρώνουν θεσμούς εντός αυτού του σώματος. Δηλαδή κάνουν τα πάντα χωρίς να ερωτηθούν προηγουμένως οι εκπρόσωποι των ε, διαφόρων αντιπροσωπιών, χωρίς να διαβουλεύονται. Και αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί μπορεί κανείς να κρύβεται πάντοτε πίσω από διαφόρους ε, παραγράφους ή μπορεί να αναφέρεται σε κάποια δικαιώματα, για παράδειγμα στον αριθμό των απολογιών που έχουν υποβληθεί. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θεωρώ αναγκαίο είναι προηγουμένως να γίνονται κανονικά οι διαβουλεύσεις. Άρα εμείς διαμαρτυρόμαστε ως πολιτική ομάδα κατά αυτού του τρόπου το οποίο πραγματικά ακυρώνει το κοινοβούλιο και παρακάμπτει τα δικαιώματά μας γίνεται τροχοπέδι στο έργο μας. Εκατομμύρια ανθρώπων, εκατομμύρια ανθρώπων ε, περιμένουν τι θα κάνουμε σήμερα. Και εσείς ε, θα το βάζετε στην άκρη. Εάν θέλετε να εκπροσωπήσετε τις πολίτες από τους οποίους, έχουμε, εκπροσωπούμε και από τους οποίους έχουμε εκλεγεί, τότε ε, θα πρέπει να ακούσετε την ε, φωνή του Κοινοβουλίου. Και εμείς ε, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το γεγονός ότι ο μεγάλος ε, συνασπισμός εδώ στο Κοινοβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει. Γιατί πραγματικά αυτό είναι απολέτος απαράδεκτο και αναξιοπρεπές. Παρακόλληση του έργου του σώματος, με το οποίο δεν συμφωνούμε. Μια ε, διαδικαστική παρατήρηση για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, για την έκθεση της ε, έκθεσης Λάγκε. Έχουν υποβληθεί 116 τροπολογίες, 87 αιτήματα για ψηφοφορίες, διαγνωστικές ψηφοφορίες και 10 για δημοτικές ψηφοφορίες. Βάσει του άρθρου 175 του κανονισμού ο Πρόεδρος ε, Σούλτ, αφού ζήτησε με τον πρόεδρο τη Αρμόδια Επιτροπή για το Διεθνέ Εμπόριο, ζήτησε από την Επιτροπή αυτή να συνέλθει για να εξετάσει τι ε, ε, τροπολογίε και τα αιτήματα αυτά. Οπότε έχει αναβληθεί η ψηφοφορία. Τώρα συζητούμε περί της συζήτησης. Εάν θα διεξαχθεί ή όχι η συζήτηση και όχι η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία έχει αναβληθεί βάσει του άρθρου 175 του κανονισμού βάσει απόφασης του Προέδρου. Ο λόγος στον Πρόεδρο Πιτέλα. Πρόεδρε Ταγιάννη, με προλάβατε. Σε πρώτη φάση στη συζήτηση αυτή δεν ήταν σαφέ αν θα αναβληθεί η ψηφοφορία ή η συζήτηση αυτή καθεαυτή. Πολύ σωστά το αποσαφηνίσατε. Δεν συζητούμε τώρα το αν θα ψηφίσουμε ή όχι. Η ψηφοφορία έχει αναβληθεί. Έχει ληφθεί απόφαση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίο αποφάσισε να αναβληθεί επειδή υπήρχαν πάρα πολλέ τροπολογίε. Το ψήφισμα αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή. Εμείς εκφράζουμε την εκτίμησή μας για την σύνεση του Προέδρου Σούλτ. το πρόβλημα του Κοινοβουλίου με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα του Κοινοβουλίου δεν είναι να επιδειχθεί αλλά να αποφασίσει δημοκρατικά. Θέλουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ε, να δείξουμε ότι αποφασίζουμε με βάση δημοκρατικά κριτήρια. Υπάρχει πραγματικό κίνδυνο να μην υπάρξει ψήφισμα. Καλά έκανε ο πρόεδρο Σούλτ. Έκανε πολύ καλά και ε, θέλει να προσπιστεί αυτό το κοινοβούλιο. Τελεία. Και έπειτα, για την συζήτηση αυτή καθεαυτή. Εμεί δεν είμαστε υπέρ κατά. Συζήτηση μπορεί είτε να γίνει είτε να συνδυαστεί με την ψηφοφορία όταν θα γίνει αυτή. Όμως το θέμα τώρα δεν είναι το θέμα ουσίας. Το ε, θεμελιώδες ζήτημα είναι ότι επειδή συμφώνησαν οι ομάδες, όχι μόνο οι ομάδες πλειοψηφίας, αλλά όλες οι ομάδες για ένα ψήφισμα, τότε ο πρόεδρος Σούλτς σωστά αποφάσισε να αναπέμψει την έκθεση και την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή. Ο κύριος Αγαπητοί συνάδελφοι, ποιο είναι αυτό το κοινοβούλιο όπου ο πρόεδρος αποφασίζει να χειραγωγήσει τον κανονισμό γιατί φοβάται ότι δεν θα πετύχει πλειοψηφία. Γιατί φοβάται ότι δεν θα πετύχει πλειοψηφία για το σύστημα διαιτησίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεξιά φιλελεύθερη πιστεύει ότι μπορεί να αποφασίσει από μόνη της για θέματα τα οποία ενδιαφέρουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο πολύ. Ποιο είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φοβάται την ψηφοφορία, που φοβάται τη συζήτηση, που φοβάται τους Ευρωπαίους πολίτες. Να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε. Ο κύριος Βέμπερ. Κύριε Βέμπερ. συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι, για, τόσο πρωί, ε, για τόσο πρωί πραγματικά είναι έντονη συζήτηση. Είναι, και θα ήθελα να διευκρινίσω και πάλι ότι είναι καθοριστικό για το θέμα κατά πόσο θα γίνει σήμερα συζήτηση ή όχι. Θα, την απόφαση θα την πάρει η Ολομέλεια. Είμαστε εμείς οι βουλευτές που θα πάρουμε αυτή την απόφαση. Λοιπόν, ε, άρα η διαδικασία είναι σωστή. Τώρα, αυτό το οποίο αποφάσισε ο Σούλτ ε, βάσει του κανονισμού και οι κανόνε είναι, είναι, ε, είναι ξεκάθαροι όταν η Ολομέλεια είναι φορτωμένη γιατί έχουν υποβληθεί πάρα πολλέ τροπολογίε, έχει το δικαίωμα να αναβάλει την ψηφοφορία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τον στηρίξουμε ώστε να διεξαχθεί σωστά το έργο του Κοινοβουλίου. Τρίτον, ε, και εγώ μπορώ να πω από πολιτική άποψη ότι φοβούμαι όταν βλέπω ότι τα δύο άκρα εδώ του σώματος, η ακροδεξιά και η ακροαριστερά, ε, υψώνουν τους ε, τόνους. Πραγματικά ανησυχώ πάρα πολύ. Ε, Κυρία Χάρμς, τελευταία παρέμβαση. Honorable you have the floor. Herr äh- θεωρώ ότι αυτή την τελευταία κατηγορία πραγματικά θα έπρεπε να τη σκεφτείτε και πάλι γιατί ο καθένας γιατί εάν ο καθένας κύριε Βέμπερ παρακαλώ ακούστε με αξιότιμοι συνάδελφοι εάν ο καθένας ο οποίος ε, ασκεί κριτική έναντι των, ε, της ιδιωτικής ε, διατησίας στο πλαίσιο της TTIP κατηγορείται ως ακροδεξιός ή ακροαριστερός και στυλιτεύεται. Διερωτώ με πραγματικά ποια είναι η ακροαριστερος και στυλιτευεται διαρωτω με πραγματικα συνεργασίας σε αυτό το σώμα. Δεν είναι το να καθόμαστε στο σκαμνί του κατηγορούμενου γι' αυτό. Ωραία λοιπόν εδώ βρίσκονται πάρα πολλοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα σε αυτή την πλευρά, αλλά και σε εκείνη την πλευρά, οι οποίοι στην εκλογική εκστρατεία υποσχέθηκαν στους ψηφοφόρους τους ότι αυτά τα ιδιωτικά δικαστήρια διαιτησίες δεν πρόκειται να συσταθούν. Και πραγματικά έχουν γίνει αυτές οι εξαγγελίες και ο Μάρτιν Σούλτς αναβάλλει την ψηφοφορία στη βάση του κανονισμού τίθεται η αναβολή αυτής της ψηφοφορίας γιατί πλέον δεν είναι ξεκάθαρο πώς η δική του πολιτική ομάδα, δηλαδή οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, πώς θα σταθούν στο, στο ύψος των προεκλογικών τους εξαγγελιών και υποσχέσεων. Και παρακαλώ, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Βιτέλα, Επιτέλα, συγγνώμη. Κύριε Επιτέλα. Κύριε Κυρία Χάρμς, δεν έχουμε συζητήσει. Εμείς παλέψαμε να υπάρχουν πάνω από 200 τροπολογίες. Το γεγονό ότι η πρόταση της κυρίας Μάιλστρομ δεν ακούγεται πλέον η ομιλήτρια. Κυρία Χάρμς, Sit down, please. Παρακαλώ καθίστε. Ο λόγος στον κύριο Καμάλ. Καθίστε παρακαλώ. Dobbiamo tolto la togliamo la parola. Onorevole. Sit down please. Καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Πώς είστε. Θα, έρθω σε σε λίγο όταν έρθει η σειρά σας. Περιμένετε. Λοιπόν, να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Επειδή όμως ελήφθη μία απόφαση με τρόπο που ελήφθη από την αριστερά, δεν θα ψηφίσουμε σήμερα. Εμείς νομίζαμε ότι είχαμε συμφωνία. Άλλη συμφωνία αυτή δεν ίσχυσε τελικά. Τώρα όμως συζητάμε κατά πόσο, όχι αν θα ψηφίσουμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα ψηφίσουμε, συζητάμε κατά πόσο θα διεξαχθεί η συζήτηση. Περί αυτού πρόκειται. Αυτοί που νοιάζονται θέλουν τη συζήτηση. Και είναι σωστό βέβαια να συζητήσουμε την ίδια μέρα που θα έχουμε και την ψηφοφορία. μπορείτε να ενθουσιάζεστε όσο θέλετε. Το θέμα είναι ότι είναι πιο σωστό να συζητήσουμε τη μέρα της προφορίας. Ακούω τους πράσινους σοσιαλιστές να συζητούν μεταξύ τους φιλικά εντό αγωγικών. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τον, τη διαδικασία αυτή η διαιτησία σε διεθνές επίπεδα. Από ό,τι φαίνεται χρειάζεται και εδώ, στην αριστερά. The The ο Τελευταίος ο κύριος Σκόβουρ από την ε, EFTD. Και μετά θα ψηφίσουμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό περιμένουν οι πολίτες. Οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση. Πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβάλει αιτήματα για να ασχοληθούμε με αυτή τη συμφωνία. Τηλεφωνήματα, email, ο καθένας και καθεμιά από εμά εδώ στο Κοινοβούλιο γνωρίζει ότι οι άνθρωποι ανησυχούν για το ζήτημα αυτό. Τι κάνουμε ακριβώς σήμερα το πρωί. Έχει προγραμματιστεί συζήτηση για το TTIP. Εάν όχι, τι θα κάνουμε, να πάμε πίσω στα γραφεία μας ή θα κάνουμε αυτό που περιμένουν οι πολίτες να κάνουμε, ε, να γίνει η συζήτηση. Η επιλογή εδώ κυρίες και κύριοι είναι επιλογή μεταξύ δημοκρατίας και ε, του να ακούσουμε το τι λένε οι πολίτες. Ή να πάμε πίσω και να κάνουμε τα πράγματα στα παρασκήνια, όπως συνήθως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή σήμερα. Αυτό περιμένουν όλοι από εμά. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, ολόκληρης της Ευρώπη Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω απολύτως με όσους τοποθετήθηκαν σήμερα το πρωί και είπαν ακριβώς αυτό που αισθάνονται και οι πολίτες. Είμαστε κοινοβούλιο γραφειοκρατών όποτε βολεύει και ένα κοινοβούλιο με μπλαμπλά και φλιαρίες όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Είναι επονίδιστο αυτό. Μόνο όταν μας βολεύει αλλάζει η κατάσταση. Αυτοί που βρίσκονται στην κεντρική πτέρυγα, οι οποίοι έχουν ε, προσκοληθεί σε μια παλιά ιδεολογία δεξιάς και αριστεράς και τέτοιων διαχωρισμών, δεν ενδιαφέρει αυτό του πραγματικούς πολίτες. Περιμένουν την ε, ε, σωστή κρίση μας και όχι τις διακρίσεις επικρίσει αριστερά και δεξιά. Κύριε Βέμπερ, σήμερα την κοινή λογική την δείχνουν οι ομάδε που βρίσκονται σε αυτή την πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Όχι εσεί που είστε στο κέντρο. Είναι σαφή η ώρα της συζήτηση. όλοι τοποθετήθηκαν, οπότε τώρα θέτω σε ψηφοφορία ηλεκτρονική. Η, η, τοποθετήθηκε. Και μάλιστα διαμακρών. Τώρα θα ψηφίσουμε, όχι, όχι. Όχι. Θέτω σε ψηφοφορία την πρόταση. Την πρόταση αναβολής της έκθεσης Λάγκε διονομαστικής ψηφοφορίας. Θέτω σε ψηφοφορία και το επαναλαμβάνω την πρόταση αναβολής. Υπέρ, όποιος ψηφίσει ναι είναι υπέρ της αναβολής. Όποιος ψηφίσει κατά είναι υπέρ του να γίνει η συζήτηση αμέσως βάσει του άρθρου 175 του εσωτερικού κανονισμού. Ο πρόεδρος αποφάσισε να αναβληθεί η ψηφοφορία. Σε αυτή τη φάση ψηφίζεται μόνον το αν θα αναβληθεί ή όχι η συζήτηση. Δεν θα γίνει ψηφοφορία ούτως ή άλλως για την έκθεση αυτή. Διονομαστική ψηφοφορίας λοιπόν. Άρχεται. La votazione è chiusa. Η ημερήσια διάταξη αλλάζει. Η έκθεση Λάγκε αναβάλλεται. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Μέχρι την ψηφοφορία στις 12. Sorry, the micro. May I draw your attention. Παρακαλώ να σας επισημάνω